Bene, possiamo dare inizio. Λοιπόν, ας, ξεκινήσουμε την διάσκεψη των προέδρων των πολιτικών ομάδων που είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη. Θέλω να καλωσορίσω, θέλω να, θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Βάντερ Ρομπάη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Σεύκοβιτς. Και δίνω μέσω το λόγο στον κύριο Βάντερ Ρομπάη που θα μας αναφέρει τα αποτελέσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα 24-25 Οκτωβρίου. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, πολλά θέματα συζητήθηκαν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μερικά προσχεδιασμένα από πολύ καιρό και άλλα ως ανταπόκριση σε τελευταίες εξελίξεις. Πριν από δύο εβδομάδες αυτά. Πάνω απ' όλα η σε αυτή έδειξε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας την υπαρξιακή κρίση του ευρώ και τώρα μπορούμε να αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια στις ευρύτερες οικονομικές προκλήσεις της ενίσχυσης, της ανάκαμψης και της ενδυνάμωσης της πολιτικής των εργαλείων μας για το μέλλον. Η ενίσχυση της ανάκαμψης σημαίνει πρώτο και απ' όλα τα συνοδευτικά μέτρα που συμφωνήσαμε νωρίτερα για χρηματοδότηση της οικονομίας και τα πολέμηση της ανεργίας των νέων για ενδυνάμωση της ε, διαρθρωτικής ανάπτυξης για εμβάθυνση της ενίας αγοράς και για καταπολέμηση του κακερματισμού. Το πρόγραμμά μας για την ανταγωνιστικότητα με την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχιστεί. Ιδιαίτερα ουσιώδες είναι να συνεχίσουμε αποφασιστικά να καταπολεμούμε την ανεργία των νέων. Θέλουμε η πρωτοβουλία για την, ανεργία, για την απασχόληση των νέων να είναι βασικό στοιχείο και μέχρι τον Ιανουάριο να έχει αρχίσει να λειτουργεί. Ήδη πέρυσι ενωσιακά κονδύλια βοήθησαν 800.000 νέους να μπουν στην αγορά εργασίας από του χρόνου με τις εθνικές εγγυήσεις της νεολαίας θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί και αναμένω ότι χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες. Πρέπει όλες οι πλευρές να εργαστούν σκληρά για να λειτουργήσει το πρώτο πρόγραμμα από το τέλος του έτους. Πολλά εξαρτώνται από το τι θα γίνει στα κράτη-μέλη και ελπίζω η διάσκεψη για την απασχόληση των νέων στο Παρίσι αυτό το μήνα να δώσει μια περαιτέρω όθηση. Η βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν ένα άλλο στοιχείο που αποφασίσαμε τον Ιούνιο. Συμφωνήσαμε να αυξήσουμε τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διπλασιάζοντας τουλάχιστον τη βοήθεια αυτή σε χώρες όπου χρειάζεται παραπάνω δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα χρήματα αυτά πρέπει να διατεθούν γρήγορα ώστε κάθε ευρώ που θα επενδυθεί να μπορεί να αποδώσει 5 ή 6 ευρώ νέων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, η απλοποίηση της νομοθεσίας θα έπρεπε να είναι επίσης ένας στόχος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Κομισιόν ήδη έχει ταυτίσει νέα βήματα για να διευκολύνει τα πράγματα ως τμήμα του προγράμματος REFIT και όλοι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να συνεχίσει και να επανερχόμαστε σε αυτό ετησίως χωρίς όμως να θυσιάσουμε τη βασική προστασία των καταναλωτών, εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Η ενδυνάμωση των εργαλείων μας για το μέλλον επίσης σημαίνει ότι πρέπει τελικά να εγκρίνουμε κατά αυτήν τη θητεία τα βασικά στοιχεία για την Τραπεζική Ένωση, μεταξύ των οποίων και ο ενιαίος μηχανισμός επίλυστος για τον οποίο το Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι υποστηρίζει την, ε, το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας που εγκρίθηκε το περασμένο μήνα θα αρχίσει να λειτουργεί σε ένα χρόνο. Ο πρόεδρος Ντράγκη μας είπε στο Συμβούλιο για τους ισολογισμούς που θα εποπτεύσει η ΕΚΤ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και οι κυβερνήσεις πρέπει να προσχεδιάσουν τα πράγματα εγκαίρως. Και εδώ είναι θέμα αξιοπιστίας. Στη συνεδρίαση τα μέλη του Συμβουλίου υποστήριξαν το θέμα αυτό και θεώρησαν ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα είναι όντως σε θέση να χρηματοδοτήσουν την οικονομική ανάκαμψη. Πέρα όμως από την Τραπεζική Ένωση πρέπει να διατηρήσουμε την ορμή για την βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση που αναφέρει η έκθεση των τεσσάρων προέδρων. Αυτή τη φορά εξετάσαμε τρόπους να ενδυναμωθεί ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα της ε, κοινωνικής διάστασης της, της Νομισματικής Ένωσης, ώστε να λάβουμε υπόψη μας περισσότερο και καλύτερα, πληρέστερα, τη κοινωνική πολιτική και την, ανυπλο... και ανεργία. Επί... Μέχρι το Δεκέμβριο θα συνεχίσει αυτή η ανάλυση και τότε θα πάρουμε αποφάσεις για τους απαραίτητους μηχανισμούς αλληλεγγύης. Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης πρόσεξε ιδιαίτερα το θέμα της ε, διαρθρωτικής ανάπτυξης σύμφωνα και με το πρόγραμμα των, της ανταγωνιστικότητας. Μετά από τη συζήτηση του θέματος της ενεργείας τον Μάιο και πριν συζητηθεί το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο, αυτή τη φορά συζητήσαμε ένα άλλο ουσιώδες θέμα, την ψηφιακή οικονομία και την καινοτομία. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί για την ενιαία αγορά πρέπει να γίνει ψηφιακή. Προ στιγμή είναι ακόμη κατακαιρματισμένοι και οι υποδομές μας απαρχαιωμένες. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη τους ειδικού που χρειάζονται για την ηλεκτρονική οικονομία. Γι' αυτό αποφασίσαμε τρία πράγματα. Πρώτον, επένδυση στην ψηφιακή οικονομία, ιδιαίτερα στι καινοτόμε υποδομέ. Δεύτερον, προώθηση μίας ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέχρι το 2015 που να είναι φιλική προς τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια εξαρτάται από δημοθετικές προτάσεις όπως η ή τα ταύτιση ή τα λογαριασμοί και ή τα πληρωμές ώστε να μπορούν να εγκριθούν πριν λήξει η θητεία. Και τρίτον, η ηλεκτρονική και ψηφιακή παιδεία Μέχρι το 2015 θα δημιουργηθούν 900.000 θέσεις ψηφιακών ε, για ψηφιακή απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση που αφορά και την κοινωνική και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σχετικά με αυτό είναι και η καινοτομία με βάση τη στρατηγική προσέγγιση που εγκρίναμε το 2011. Γενικά λοιπόν αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία που έχει μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν στην Ένωση να επιτρέψει στην ηγετική θέση που είχε στην ψηφιακή καινοτομία πριν από 20 χρόνια και την οποία έχει χάσει. Όπως στον τομέα της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών και η ενιαία αγορά έχει κατακαιρματιστεί στα ψηφιακά θέματα και στις τηλεπικοινωνίες. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα για απασχόληση και ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης ασχολήθηκε με πρόσφατα ανησυχητικά ή τραγικά γεγονότα. Όλοι έχουν σοκαριστεί από αυτά που έγιναν κοντά στη Λαμπεντούζα. Όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να αναλυφθεί κάποια αποφασιστική δράση για να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Με τρεις αρχές πρόληψη, προστασία και αλληλεγγύη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να συζητούμε τις ρίζες της παράνομης μετανάστευσης σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης. Πράγμα που συμπεριλαμβάνει και αναπτυξιακή βοήθεια καθώς και περισσότερο διάλογο με αυτές τις τρίτες χώρες. Καταπολέμηση της δουλεμπορίας και αυτό και στις δικές μας χώρες και στις χώρες προέλευσης. Για την προστασία της ζωής ζητήσαμε σύντομη, γρήγορη, αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων Eurosur, γιατί έτσι θα σωθούν πολλές ζωές. Ζητήσαμε δυνάμωση της δράσης του Frontex στη Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ένωσης. Πέρα από αυτό συμφωνήσαμε όλοι ότι είναι ουσιώδες και επίγον να δούμε τι μπορεί να γίνει βράχη πρόθεσμα. Γι' αυτό ζητήσαμε από την καινούργια αυτή task force για τη Μεσόγειο, τη οποία ηγείται η Κομισιόν, μαζί με τη διπλωματική υπηρεσία των διαφόρων χωρών, να υποβάλουν σύντομα προτάσεις για πιο αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εργαλείων. Οι μεταναστευτικές ροές είναι πολύπλοκα φαινόμενα και πρέπει να τα σκεφτούμε καλά όταν θα συζητήσουμε ευρύτερα το μέλλον των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης τον Ιούνιο του 2014. Κυρίες και κύριοι, όπως λέει και ο τύπος, συζητήσαμε και για τις τελευταίες εξελίξεις για τα θέματα της κατασκοπίας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, ανησυχούν και την ανησυχία αυτή την ε, είδαμε και στις συζητήσεις μας. Είναι κατανοητή αυτή η ανησυχία. Γιατί μια εταιρική σχέση όπως μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη και για τις μυστικές υπηρεσίες και ως προς τις μυστικές υπηρεσίες. Αν λείπει η εμπιστοσύνη μπορεί να καταστραφεί η συνεργασία στο θέμα της συλλογή πληροφοριών, τομέας που όπως όλοι ξέρουμε είναι πολύ ουσιαστικό για την καταπολέμηση της τορομοκρατίας. Σε μια κοινή δήλωση οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων σημείωσαν την πρόθεση της Γερμανίας και της Γαλλίας να έχουν διμερείς συνεννοήσεις με τη ΣΥΠΑ για να βρεθεί πριν το τέλος του χρόνου μία κατανόηση για το θέμα των αμοιβαίων σχέσεων στο θέμα της συλλογή πληροφοριών και για τη δημιουργία περισσότερης αφήνειας ως προς το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συλλέγουν τις πληροφορίες αυτές. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να συνδυάσουν, με αυτές τις ζητήσεις, αλλά προς στιγμή θέλουμε να δούμε αν και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η πρωτοβουλία. Δεν είναι η μόνη. Μετά από τις κατηγορίες περί του πρίσμα τον Ιούλιο, μια ομάδα εργασίας Ένωσης είπα για τα θέματα αυτά, θα αναφέρει τα αποτελέσματά της πριν λήξει το έτος. Είμαι πεπισμένος ότι οι πρόεδροι και πρωθυπουργοί της Ένωσης στην κοινή αυτή δήλωση έδωσαν ένα στεναρό μήνυμα προς τη ΣΥΠΑ ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και ότι αναμένουμε από αυτές τις ΗΠΑ να το προσέξουν ιδιαιτέρως. Κυρίες και κύριοι, τέλος προετοιμάσαμε και τη διάσκεψη του Βίλνιους με τους έξι ανατολικούς μας εταίρους που θα γίνει σε τρεις εβδομάδες. Ελπίζουμε να ληφθούν εκεί σημαντικές αποφάσεις ιδιαίτερα ως προς την Ουκρανία εάν υπάρξει απτή πρόοδος για το σεβασμό των όρων που είχε θέσει τον περασμένο Δεκέμβριο ήδη το Συμβούλιο Εξωτερικών. Η Ουκρανική ηγεσία ξέρει τι πρέπει να γίνει και η Συμφωνία Σύνδεσης θα είναι μια δοκιμή για όλους τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης παρόμοιες συμφωνίες είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε με τη Μολδαβία και τη Γεωργία που να υπογραφούν το επόμενο φθινόπωρο. Γενικά λοιπόν ήταν ένα πολύ φορτωμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συζήτησε πολλά θέματα κλειδιά και έπαιξε πλήρω το ρόλο του στρατηγική κατεύθυνση, δημιουργία στρατηγική κατεύθυνση τη Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Βαν Το λόγο έχει τώρα ο Αντιπρόεδρος κ. Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρίε και κύριοι κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος Μπαρόζο δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρόν εδώ γιατί είχε υποχρεώσεις εκτός ε, Βρυξελών, αλλά θέλει να μοιραστεί μαζί σας τις απόψεις της Επιτροπής για την πρόσφατη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως ήδη ανέφερε και επανέλαβε ο κύριος Βαν το Συμβούλιο κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την ψηφιακή οικονομία και την κοινοτομία, την οικονομική κατάσταση, την εμβάθμιση, την εμβάθυνση της ε, ΟΝΕ, την μετανάστευση, την ε, ανατολική συνεργασία και τις δραστηριότητες αντικατασκοπίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, για την εξαιρετική παρέμβασή του και την επικοδομητική προσέγγιση του στην ε, σύνηθη παρουσίασή του στο ξεκίνημα του Συμβουλίου. Ιδίω δε ε, το αίτημα του να ζητηθεί ταχεία ολοκλήρωση των νομοθετικών εκκρεμωτήτων πριν τις εκλογές. Βασικό στόχο μα θα είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο, την ε, νομοθεσία για τις εταιρείες και τους προϋπολογισμούς για το 2013 και 2014. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε μια ζωηρή και ε, σημαντική συζήτηση για την ψηφιακή οικονομία. Η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο γίνεται τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία που προκύπτει, ε, που δεν επιτυγχάνεται λόγω της, του κατακαιρματισμού της αγοράς και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μέτρα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για να υιοθετηθούν όλες οι αναγκαίες αλλαγές, καθώς και να παροτρύνει και να προωθήσει την, την επένδυση καινοτομία δημοσίων και ιδιωτικών πόρων. Η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς το 2015 είναι λοιπόν σημαντική προτεραιότητα για μας και ελπίζουμε στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει ταχεία πρόοδος για να υιοθετηθούν και τα πακέτα για τις ε, τηλεπικοινωνίες και η βασική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων πριν τις ευρωεκλογέ. Ο πρόεδρος Μπαρόζο πίεσε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν το έργο τους στην εγγύηση για τους νέους και την πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση των νέων. Είναι αναγκαίο να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη έγκαιρα τα, σχέδια, τα σχετικά σχέδια πριν το τέλος του έτους για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ταχύτερου δυνατό. Αυτό θα είναι σημαντικό και για να εξασφαλιστεί ότι τα 6 δις ευρώ για την πρωτοβουλία απασχόλησης νέων θα δαπανηθούν όπως πρέπει. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να τα βοηθήσει να προετοιμάσουν τα σχέδια. για την ανάπτυξη θα αναλύσει όλα αυτά τα θέματα σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Καλωσορίζουμε την υποστήριξη της στην αύξηση του επίπεδου δεσμεύσεων για την υλοποίηση των οικονομικών, πολιτικών και τι μεταρρυθμίσει που προκύπτουν από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Προ τα πλαίσια αυτό, ο Πρόεδρο Μπαρόζο υπογράμμισε εκ νέου ότι τα πρώτα βήματα για την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών θα πρέπει να στηρίζονται και στην, οικονομική, και στην κοινοτική μέθοδο και στο εξάμεινο. Κατόπιν εξετάσαμε την Τραπεζική Ένωση. Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι, ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρξει συμφωνία επί της Γενικής Προσέγγισης για τον ενιαίο μηχανισμό απόσβεσεων και έχουμε επίγνωση ότι η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί, είναι δύσκολη, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την ε, δυνατότητα αυτή. Ο πρόεδρος Μπαρόζο επιβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί ούτως ώστε ο μηχανισμός αυτός να ολοκληρωθεί πριν τις ευρωεκλογέ και η σχετική νομοθεσία για την, ε, τις εγγυήσεις και την, ε, και την ε, απόσβεση των τραπεζών μέσα στο έτος. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει στην συνολική αξιολόγηση των ισολογισμών των τραπεζών, κάτι που θα είναι βασικό στοιχείο για το τραπεζικό σύστημα της Ένωσης. Έγινε μια πρώτη σημαντική συζήτηση μεταξύ αρχικών κρατών και κυβερνήσεων για τις προτάσεις της Επιτροπής να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Η πρόταση της Επιτροπής ε, για την ε, κοινή έκθεση, για το βαθμολόγιο, περιλάβαν μια σειρά διατάξεων που ε, κρίθηκαν θετικές. Ταυτόχρονα κατέστη προφανές από τη ζητήσεις ότι συνέχιζαν να υπάρχουν διαφορετικές ευαισθητησίες και τα, μέσα, τα βασικά εργαλεία δράσης στον τομέα αυτό εξαρτώνται ακόμα από τα κράτη-μέλη. Με ικανοποίηση είδαμε επίση ότι η πρόταση της Επιτροπής για το REFIT ήταν ευπρόσδεκτη που επιτρέπει να, προσαρμόσει τη μελλοντική δραστηριοποίησή μας για την αξιολόγηση και διαμόρφωση, το, αξιολόγηση των παλαιών προτάσεων και διαμόρφωση νέων προτάσεων. Ε, να ευχαριστήσω ε, και τον κύριο Σούλτς για την προσωπική υποστήριξη του. Ήταν ένα, το ρεύτη ένα καλό πρόγραμμα για μια πιο ορθολογική, απλή και λιγότερο γραφειοκρατική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ήταν ωστόσο σαφές ότι το ΡΕΦΤ είχε στόχο να μειώσει τον ε, το διοικητικό φόρτο τους πολίτες και τις ε, εταιρείε, αλλά να μην μειώσει την κοινοτική ρύθμιση στους τομείς προστασίας ε, των εργαζομένων, των καταναλωτών και των ε, πολιτών. Ούτε να μειώσει τα επίπεδα προστασίας. Στο πλαίσιο της πρόσφατης τραγωδίας στην Λαμπεντούζα το Συμβούλιο συζήτησε τα μεταναστευ... τις μεταναστευτικές ζωές και είναι σαφές ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να συνδιαλέξουμε ανθρωπιστική αντα... Ε, την ανθρωπιστική ε, ανταπόκριση με τις επιταγές ασφάλειας. Η Ένωση θα προσπαθήσει να βελτιώσει, τους τομείς σε διάφο... Ε, να βελτιώσει κατάσταση σε διάφορους τομείς όπως την διάσωση στη θάλασσα και την ενίσχυση των χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες, να βελτιώσει την καλύτερη συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης για να καταμολεμήσει μεταξύ την διακίνηση ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα. Η δημιουργία μια task force τη Επιτροπή ήταν εξαιρετικά πρόσδεκτη και περιμένουμε πολλά πράγματα τι επόμενε εβδομάδε. Ήδη θα συζητήσει το θέμα αυτό το Συμβούλιο εκ νέου τον Δεκέμβριο. Ο πρόεδρο Βαν Πόρε αναφέρθηκε και στην Σύνοδο Κορυφή με, του Ανατολικού με του ανατολικού γείτονέ μα στο Βίλνιο. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για τη βελτίωση των σχέσεων προς την ανατολική γειτονιά μας, ε, παρέχοντας την Ουκρανία και άλλες χώρες, εφόσον οι χώρες αυτές μάλλον τηρούν τις προϋποθέσεις που θέσαμε. Η συμφωνία σύνδεσης και μια ε, συμφωνία, σημαντική συμφωνία συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί με την ε, Ουκρανία, ενώ να μονογραφηθούν αντίστοιχε συμφωνίες με τη Μολδαβία. Επίσης έγιναν συζητήσεις για τις πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της κατασκοπίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν έρθει σε διμερείς επαφής με τις ΗΠΑ για να καταλάβουν καλύτερα την κατάσταση με αυτό. Όπως σας είπα, η μερίσια διάταξη του Συμβουλίου ήταν πλούσια. Πιστεύω ωστόσο ότι σε πολλά από τα βασικά ζητήματα επιτέχθηκε πραγματική πρόοδος και ήταν καλό πλαίσιο για τις περαιτέρω δραστηριότητες ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκέμβριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε.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 Κύριε Αντιπρόεδρε, τέθησαν διάφορα θέματα που στηρίζουμε και τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και να ενισχύσουμε τις οικονομίες και να προσφέρουμε θέσεις απασχόλησης στους ε, πολίτες. Τα επίπεδα ενεργείας είναι απαράδεκτα. Χρειάζονται λοιπόν διαρθρωτικές αλλαγές ε, για να επιτύχουμε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Εμείς χαιρετίζουμε τις ενδείξεις βελτίωσης στην οικονομία μας, παράλληλα όμως γνωρίζουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Και αυτό δεν το λένε μόνο τα στοιχεία, εδώ μιλάμε για θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες. Υποθέτουμε ότι έγινε κάποια πρόοδος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά παραμένουμε ακόμα ανήσυχοι για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις ε, προτεραιότητές της. Εμείς πιστεύουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα πρέπει να συνεχιστεί ο συντονισμός των ε, δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών ε, αυτά που επηρεάζουν το κεφάλαιο σε μια χώρα επηρεάζουν και σε άλλη. Το μάθημα λοιπόν από την οικονομική κρίση είναι ότι σήμερα είμαστε τόσο αλληλένδετοι που πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να λειτουργούν οι οικονομίες μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει κατά κάποιο τρόπο αυτό. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί η ε, Τραπεζική Ένωση. Μια κακή εισαγωγικά τράπεζα δεν θα μπορεί πλέον να αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει επιγόντως να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση πριν από το τέλος της νομοθετικής περίοδου. Στην ΕΚΤ έχουμε δώσει την εντολή να εποπτεύει τις τράπεζές μας. Αυτό όμως είναι μόνο το πρώτο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε με έναν ενιαίο ε, μηχανισμό διάσωσης ε, και όλο αυτό να ολοκληρωθεί ε, πριν από το τέλος της θητείας μας. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η Τραπεζική Ένωση μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνο εάν ε, στηριχθεί στις ενέργειές της. Εμείς καλούμε το Συμβούλιο να αποφασίσει το ταχύτερο δυνατόν για τα περίφημα backstops, διότι η αξιοπιστία ε, βρίσκεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να παραμείνουμε φιλόδοξοι όσον αφορά γενικότερα την ανάκαμψη της οικονομίας. Χρειαζόμαστε περισσότερο θέσεις απασχόλησης από οτιδήποτε άλλο. Ανταγωνιστικότητα, όχι αύξηση της φορολογικής βάσης, διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να ευημερήσουν οι μικρομεσαίες και να προσφέρουν θέσεις απασχόλησης. Να αρθούν οι φραγμοί, να εμβαθυνθεί η εσωτερική αγορά Αυτά βοηθούν στο να επιτύχουμε το στόχο μας. Γι' αυτό λοιπόν το ΕΛΚ στηρίζει ανεπιφυλακτά την έκκληση του Συμβουλίου να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να ελαφρυνθεί το βάρος της ε, νομοθεσίας κυρίως για τις ΜΜΕ γιατί αυτές είναι η κινητήρια δύναμη των θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης. Πρόεδρε, πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι στην εφαρμογή του διπλού και του εξαπλού πακέτου εμείς ε, δεν θα ενδώσουμε. Ε, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η νέα οικονομική διακυβέρνηση θα διαθούν και πάλι ένα αμφιβόλο. Εάν λοιπόν η διαδικασία μεταρρυθμίσεων επιβραδυνθεί, όχι μόνο θα χάσουμε από ενθουσιασμό, αλλά σιγά σιγά θα διολυστήσουμε και στην κρίση από την οποία αγωνιζόμαστε να ξεφύγουμε. Τα τελευταία στατιστικά δεδομένα από την Ιρλανδία δείχνουν ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα με φιλόδοξες ε, μεταρρυθμίσεις, οδηγούν σε αποτέλεσμα και θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση. Επίσης χαιρόμαστε για το ότι το Συμβούλιο επιτέλους κατόρθωσε να βρει τα χρήματα που έλειπαν για το 2013. Εκπλησόμεθα μόνο που χρειάστηκε τόσο πολύ καιρό. Ήδη τον Ιούλιο ήμασταν πεπισμένοι ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία. Το Κοινοβουλίο ήταν απόλυτα σαφέ τα βασικά του αιτήματα. Πρώτον, τα 3,9 δις για το 2013 ε, πρέπει να καταβληθούν και δεύτερον να ζητήσουμε μια ρήτρα διάσωσης και επίσης να συσταθεί ομάδα υψηλού επίπεδου για να εξετάσει το σύστημά μας των ιδίων πόρων. Αυτά ήταν λογικά αιτήματα και πιστεύουμε ότι είχαν ήδη γίνει αποδεκτά. Και πρόεδρε, τα 3,9 δις ε, δεν είναι ε, ένα νέο αιτήμα, νέα χρήματα, αλλά είναι χρήματα τα οποία τα κράτη-μέλη που τα μπλοκάρουν τώρα τα έχουν ήδη δαπανίσει σε προγράμματα όπως το Έρασμος, όπου 250.000 ε, νέοι κάθε χρόνο μπορούν να υποφεληθούν από πανεπιστήμια άλλης χώρας. Είναι λοιπόν χρήματα που δαπονήθηκαν σε υποδομές, νέους δρόμους, γέφυρες. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι μιλάμε για 11.000 ε, χιλιόμετρα που ανανεώθηκαν ή κατασκευάστηκαν με την τελευταία δημοσιονομική προοπτική. Επίσης χρήματα που δαπανήθηκαν στον ενεργειακό τομέα για να μην εξαρτώμεθα τόσο πολύ από τρίτους. Για δέστε λιγάκι την τραγωδία της Λαμπεντούζα. Ήταν και χρήματα, ίσως όχι αρκετά, για τη Frontex, ε, για να παραμείνουν τα ε, σύνορά μας ασφαλή. Όλα αυτά τα ζήτησε το Κοινοβούλιο και εξακολουθεί να τα ζητάει και ζητάει να πληρωθούν οι λογαριασμοί όταν θα κατατεθούν γιατί αυτές και άλλες κοινέ δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα ωφελήσουν τους πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο λόγος που επανέλθουμε στο θέμα αυτό ε, και γιατί το ζητάμε να παραμείνουν σε τάξη τα οικονομικά μας είναι γιατί ανησυχούμε. Αφενός επιμένουμε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να περικοπεί ενώ παράλληλα ζητάμε περισσότερες ευρωπαϊκές δράσεις. Ε, Παραδείγματος χάρη μετανάστευση που αναφέρθηκα. Πρόεδρε, ε, ας δείξουμε μια ματιά στο τι συζητάμε σήμερα ε, και τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνοβούλιο. Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τι θέλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν η Ένωση να επενδύσει σε καινοτομίες, να προάγει μια ενιαία ψηφιακή τηλεπικοινωνιακή αγορά και θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα πάντα για να ολοκληρωθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά το 2013. Το στηρίζουμε αυτό ανεπιφύλακτα γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι αυτές οι επενδύσεις προσελκύουν ιδιωτικές, ε, τον ιδιωτικό τομέα και έτσι πενταπλασιάζουν τα χρήματα που έχουν επενδυθεί. Ως ομάδα ανέκαθεν ισχυριζόμασταν ότι οι κοινέ επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην προαγωγή νέων ε, δεξιοτήτων στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι απαραίτητα. Λέμε όμως επίσης ότι αν θέλουμε θέσεις απασχόλησης με μηδενικό κόστος, τότε η κοινή αγορά είναι ο μόνος ε, πραγματικός ε, δρόμος. Και η ψηφιακή ενιαία κοινή αγορά κυρίως ε, προσφέρει τεράστιο δυναμικό. Σε αυτόν τον τομέα θα υπάρξουν 900.000 ε, κενά μέχρι το 2014. Θέλουμε λοιπόν κοινέ ενέργειες σε αυτόν τον τομέα. Και κυρίως ε, πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε σταθερά αλλά και σε κινητά δίκτυα. Γι' αυτό μιλάμε για το ε, σχετικό πρόγραμμα. Η δική μας η ομάδα στηρίζει την πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων ε, και ε, για εγγύσεις για τους νέους. Συζητήθηκε αυτό στο Συμβούλιο. Η προτεραιότητά μας εξακολουθεί να είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ απλά. Ως κοινωνία δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αν το 50% των νέων μας είναι άνεργοι. Πρόεδρε, η Ευρώπη δεν είναι ήπειρος ε, με πλουτοπαραγωγικές πηγές. Γι' αυτό να δώσουμε έμφαση σε δεξιότητες, εκπαίδευση, διαβιωμάθηση και κινητικότητα. Ανέκαθεν τα λέγαμε αυτά στο Κοινοβούλιο και αυτά ψηφίσαμε τον Οκτώβρη για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που έπρεπε να γίνει πριν από πολύ καιρό. Πρόεδρε Βαν Οχομπέι, εγώ ανησυχώ για το ποιο τελικά θα πληρώσει για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες αν όχι το ευρωπαϊκός προπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μα ε, μας ανησυχεί το υπάρχει αυτό, αυτή η στασιμότητα, το διέξοδο σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ε, μοιάζει να υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες για την Ευρώπη, όμως κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ε, οικονομική ευθύνη που σχετίζεται με αυτές τις πρωτοβουλίες. Δυστυχώς αυτά σημαίνουν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είτε υπόσχεται προγράμματα που ποτέ δεν θα υλοποιηθούν, είτε η ασθένεια ε, των ε, ε, δαπανών που έχει μπει στις οικονομίες μας θα μπει και στον κοινωτικό προϋπολογισμό. Κύριε Βαν Χομπέι, το δημοσιονομικό, το πολιτές πλαίσιο είναι πάνω από, δεν είναι μόνο ένα οικονομικό εργαλείο. Οι κοινωνίες καλούνται να επιδείξουν αλληλεγγύη για να βρουν κοινέ λύσεις. Η δική μας η ομάδα θα συνεχίσει να πιέζει για ισχυρή Ευρώπη. Σε όλους τους τομείς, διότι πιστεύουμε ότι η συνεργασία συνεπάγεται υπεραξία αξία που, ε, <clears throat> που ωφελεί γενικά την Ευρώπη, στο σύνολό της. Ευχαριστούμε την κυρία Βόρτμαν Κόλ και τώρα ε, θέλω να δώσω το λόγο στον αξιότιμο κύριο Γκερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Δεν θα σας εκπλήξει αν σας πω ότι η ομάδα μου δεν έχει την ίδια άποψη για το τι έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι σύνηθες ε, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όταν έρχεστε να μας παρουσιάσετε τι έγινε στη συνάντηση. Πριν από χρόνια στην Ισπανία υπήρχε μια, ένα ανέκδοτο, χαζό κάπως, που έλεγε ρωτούσε κάποιος κάνει κρύο ή ζέστη και η απάντηση ήταν ούτε κρύο ούτε ζέστη, μηδέν βαθμοί. Μηδέν βαθμοί σημαίνει πάγο παντού στην Ισπανία, τη Γερμανία, τις Βρυξέλλες. Και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του Συμβουλίου. Ούτε κρύο, ούτε ζεστό. Κάποια σημαντικά μέτρα πέρασαν για το 2015, αλλά δεν υπήρξε επαρκής ισχύς για να τα εξετάσουμε και εν τέλει ούτε καν τις προσδοκίες μας δεν απογοήτευσε γιατί δεν είχαμε ψηλές προσδοκίες. Προφανώς δεν βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Το ευρώ δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Ο, ο ασθενής έφυγε από την εντατική, πήγε στην, ε, σε κλίνη, αλλά είναι άρρωστος, συνεχίζει να είναι άρρωστος. Και σιγά σιγά, αν δεν υπάρξουν μόνιμα μέτρα αποκατάστασης, θα μείνει χρόνια ασθενής. Το Συμβούλιο μπήκε σε μια ε, πορεία αυτό, ε, ικανοποίησης που λέει τα χειρότερα πέρασαν, ας ξεκουραστούμε, ας πάρουμε μια ανάσα. Δεν υπάρχει λόγος για να μένουμε τόσο ε, ικανοποιημένοι και δεν υπάρχει λόγος να, παίρνουμε, να σταματάμε. Τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία στην Ευρωζώνη, τις του τελευταίου τριμήνου που γνωρίζουμε είχαμε ανάπτυξη 0,3%. Σε αιτήσια βάση ωστόσο, αν συγκριθεί με το αντίστοιχο τρίμηνο του 12, βρισκόμαστε ακόμα στο 0,5% μείωση. Απασχόληση. 17 χώρες της Ένωσης βρίσκονται με ποσοστό ανεργίας άνω του 10%. 5 χώρες είναι άνω του 15%. 2 άνω του 20%. Σύμφωνα με συνενδική άποψη των οικονομολόγων, σε πολλές, σε πολλές από τις χώρες αυτές, η μείωση στο 10-15% θα, θα πάρει μια δεκαετία. Υπάρχουν προφανώς χώρες που είναι σε χειρότερη κατάσταση από άλλες. Η κατάσταση ωστόσο είναι σοβαρή σε όλη την Ένωση. Η φτώχεια επίσης αυξήθηκε. Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους σήμερα είναι φτωχός. Η ανισότητα αυξήθηκε σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι. Όχι. Με τον χαμηλό πληθωρισμό της Ένωσης, 0,7%, με υπερτιμημένο ευρώ, υπάρχει χώρος για μέτρα επέκτασης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Και υπάρχουν πολλές χώρες Ένωσης που δεν έχουν κρίση και θα μπορούσαν να, και θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τέτοιες πολιτικές. Ωστόσο πρέπει να προχωρήσουμε προς την Τραπεζική Ένωση. Και ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας ήταν ένα βήμα μπρο. Όλα τα άλλα θέματα που βρίσκονται ωστόσο καθοδόν και ο ενιαίος μηχανισμός εξυγένσης τραπεζών ή και το τελικό ενιαίο ταμείο εξυγένσης θα αργήσουν. Ή θα έρθουν το 2016 όπως θέλει η Επιτροπή ή το 2018 όπως θέλει το Συμβούλιο. Καμία από τις δύο ημερομηνίες δεν δίνει απαντήσεις στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κατασκοπία. Η αντίδραση του Συμβουλίου ήταν εξαιρετικά δειλή. Όλοι γνωρίζουμε τη φράση του Λόδου Πάλμερστον. Η Αγγλία δεν έχει αιώνιους φίλους, ούτε αιώνιους εχθρούς. Τα συμφέροντά της μόνο είναι αιώνια. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε μια τέτοια συμπεριφορά από πλευρά ΗΠΑ. Δεν είναι νόμιμο να παρακολουθούνται εγκαταστάσεις, οργανισμοί και υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι νόμιμο να ερευνώνται και να παρακολουθούνται ηγέτες των χωρών της Ένωσης. Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούνται πολίτες στην καθημερινή του ζωή. Αυτό είναι αδίκημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαίωμα στην προσωπική ζωή είναι θεμελιώδες δικαίωμα της Ένωσης. Η απάντηση του Συμβουλίου στο σημείο αυτό ήταν αδύναμη. Πολύ πιο ξεκάθαρη ήταν η απάντηση του Κοινοβουλίου όταν υιοθετήσαμε το ψήφισμα για το αίτημα μας για την, για την αναστολή της Συμφωνίας SWIFT. Ισχυρότερη ήταν η απάντηση του Κοινοβουλίου όταν πολλές επιτροπές, ιδίως η ΛΥΜΠΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα, μετέφερε την ενόχληση του Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα την πρόταση να υπάρξει κοινή δουλειά, κοινή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως το Κογκρέσο τον είπα, για να αντιμετωπιστούν πολυμερείς απαντήσεις, όχι μόνο διμερείς απάντηση. Να τονίσω στην δεύτερη περίπτωση να ασχοληθώ με άλλα θέματα ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την απόφαση του Συμβουλίου που ερμηνεύτηκε ότι αναβάλουμε για το 2015 το πακέτο για την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι θεμελιώδη δικαίωμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμέσω. Ούτε συμφωνούμε ώστε το θέμα της προστασία των δεδομένων να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις τη Συμφωνίας Σύνδεση Ελευθερία Εμπορία. επίπεδο της εποπτείας αλλά και στα θέματα του Ταμείου της Εξυγίανσης των Τραπεζών για να επιστρέψει κάποια ροή ρευστού στην πραγματική οικονομία. Σημειώνουμε για την Νομισματική Ένωση ότι μόνο για εμβάθυνση μιλάει ενώ όλοι ξέρουμε ότι η θεσμική λειτουργία της δεν είναι η σωστή, δηλαδή δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα, χρειάζονται νέες οργανώσεις όπως με την Τραπεζική Ένωση και κάποια δυνατότητα φορολογικών δυνατοτήτων στην Ευρωζώνη. Η κρίση δεν έχει τελειώσει και αν συνεχίσουν τα πράγματα με τον ίδιο ρυθμό και σε 20 χρόνια έτσι θα είναι τα πράγματα. Για τις μεταναστευτικές ροές λυπούμαστε για την απώλεια τόσων ζωών στα σύνορα της Ένωσης πρέπει να γίνει κάτι απτό και όχι απλώς να πούμε ότι θα αναβάλουμε τη λύση για τον Ιούνιο του 2014. Αυτό το θεωρούμε τελείως κοινικό. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι όταν σημειώθηκε μεγάλη μεταναστευτική ροή και κύμα από τη Βόρεια Αφρική λόγω της ε, πολιτικής αραβικής άνοιξης δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και ακόμη δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα υπάρχει προοπτική με περισσότερων ακόμη μεταναστευτικών ροών λόγω της, ε, του προβλήματος της Συρίας και πάλι δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Ίσως τα ίδια να γίνουν και με το Λίβανο, με τη Λιβύη και πάλι θα είμαστε απροετοίμαστοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παρβανόβα. Κυρία Ρεβέκα Χάρμς έχει το λόγο. Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, για μένα αλλά και για πάρα πολλούς άλλους πολίτες ε, πιστεύουμε, που πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές αξίες. Ε, αυτά τα τελευταία συμβούλια ήταν μια μεγάλη απογοήτευση. Παραδείγματο χάρη, αποφασίστε να μιλήσετε για τη Λαμπεντούζα, αλλά τελικά αποδείξατε δεν ήσασταν σε θέση να διορθώσετε έστω και κατά τη, την πολιτική ασύλου της Ένωσης. Δεν φροντίζουμε ούτε καν να εφαρμόσουν τα κρατημέλη ή ελλειπείς έτσι και αλλιώς κανονισμοί. Δεν έχουμε κανένα τρόπο να ασκούμε πίεση αυτή η κατάσταση στη Συρία είναι ανυπόφορη και δεν κάνουμε τίποτα και η πολιτική μας περί Αφρικής πρέπει και αυτή να συζητηθεί επιγόντως διότι έχει κάποια συγκεκριμένα αίτια και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Δεύτερο σημαντικό θέμα δικαιώματα του πολίτη, προστασία δεδομένων. Εδώ και κάποιες εβδομάδες, χάρη στον Edward Snowden, γνωρίζουμε όχι μόνο ότι γίνεται παρακολούθηση τηλεφώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ότι παρακολουθούν και το τηλέφωνο της Καγκελαρίου από τότε που αρνήθηκε να είναι ε, ουραγός των Αμερικανών ε, στον πόλεμο κατά του Ιράκ. Και τι κάνατε ή τι κάναμε, τίποτα ο κανονισμός περί προστασίας δομένων ε, μεταφέρεται σε ελληνικές ε, καλένδες. Κάπως έτσι πολύ ασαφώς ε, λαμβάνεται η απόφαση να σταλεί μια επιστολή στην Αμερική και διαβάζω στη Γερμανία ότι θα το πω πολύ καθημερινά διαβάζω ότι ο μεγαλύτερός μας ε, Ρουφιάνος, ε, κατάσκοπος με συγχωρείτε, ε, αποφασίζεται να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες απλά και μόνο για να συζητήσει με τον ομόλογό του τον αντίστοιχο υψηλότατο κατάσκοπο για το τι μπορεί να γίνει. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι στο τελευταίο Συμβούλιο απέτυχαν παταγωδός. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσαμε να ανασταλεί η συμφωνία SWIFT. Εγώ πιστεύω βέβαια προσωπικά ότι έπρεπε να ανασταλεί και η συμφωνία PNR. Το θεωρώ ότι είναι τεράστιο σκάνδαλο το ότι οι Αμερικανοί μας λένε σκέπτονται κάπως ε, να περιορίσουν τη βιομηχανική κατασκοπία. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν οι ε, διαπραγματεύσεις τι τι, αν αυτό λοιπόν δεν είναι ευρωπαϊκή αξία, ε, τότε τι είναι κυρίες και κύριοι. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα. Το γεγονός ε, ότι ξαφνικά ε, μας λένε έτσι ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις να μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως το, στο μέλλον, να υπάρχουν κάποια χρήματα να δοθούν στις χώρες κρίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ε, τα κράτη αυτά ε, θα υποταχθούν στις απόψεις της κυρίας Μέρκελ ε, για μεταρρυθμίσεις. Θέλω να μάθω πώς το βλέπει αυτό το κοινοβούλιο και θέλω να γνωρίζω ε, κατά πόσον ο κύριος Σόλτς, ο οποίος ξαφνικά στον τύπο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο αγαπημένος της μαμάς Μέρκελ, κατά πόσον ο κύριος Σούλτς θα λάβει το λόγο και να δω τι θα πει για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις αξίες της κοινή λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα έχει να πει όχι για μια απλή μεταρρύθμιση μεταρρύθμιση και λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ο κύριος Τζέφρι δεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ομάδα μας χαιρετίζει την πρόοδο που σημείωσε το Συμβούλιο για την απελευθέρωση της νομοθεσίας για τη βελτίωση των εταιρικών σχέσεων και για την ε, πληρέστερη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και στα ψηφιακά. Κατά τα άλλα, σωστά τόνισε ο πρόεδρος Μπαρόσο ότι πολλά από τα υπόλοιπα θέματα καλύτερα θα λύνονταν εθνικά. Το Μπερλεμόν γενικά φαίνεται ότι πιστεύει στην αρχή της business as usual. Από το 2003 και πάλι το 2007 είχαμε θέσει διάφορα προβλήματα τα οποία δεν ακολουθήθηκαν από καμία δράση. Γιατί τώρα τα ξανασυζητούμε. Ίσως ο Επίτροπος Κάλλας πρέπει να το ξανασκεφτεί. Γιατί ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη λύση θα ήταν να μειωθεί ο αριθμός των γραφειοκρατών και των γενικών διευθύνσεων. Λιγότερη γραφειοκρατία σημαίνει περισσότερη ανταγωνιστικότητα και μείωση του ύψους του ε, ενωσιακού προϋπολογισμού. Για το εμπόριο χαιρετίζουμε την εμπορική συμφωνία με τον Καναδά, αλλά δεν πρέπει εδώ να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας. Υπάρχει και το πρόβλημα με την Ινδία. Αυτό γιατί δεν συζητήθηκε. Γιατί μέχρι τις επόμενες εκλογές και εδώ και εκεί θα έχει λήξει η ευκαιρία αυτή για να το συζητήσουμε. Δεν πρέπει τέτοιου είδους ευκαιρίες να τις ε, παραγνωρίζουμε για τη μετανάστευση. Τα γεγονότα στη Λαμπεντούζα δείχνουν ποιο είναι το πρόβλημα των χωρών στα σύνορα της Ένωσης, αλλά δύο τρίτα των ετούντων άσυλο αφορούν μόνο πέντε βόρειες χώρες εξών και η δική μου. Το θέμα δεν είναι να δημιουργηθούν νέες μορφές νόμιμης μετανάστευσης, αλλά η πρόληψη και η αντιμετώπιση του προβλήματος στη ρίζα, του. Πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες επιστροφών με τις χώρες κυρίως της Βόρειας Αφρικής για να σταματήσει επιτέλους αυτή η ανεξέλεγκτη και μαζική μετανάστευση γιατί η θέση της Ένωσης μέχρι τώρα απλώ δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Τώρα για την κατασκοπία. Ποια είναι η πραγματική βάση για την δίθεν αυτή αγανάκτηση της Κομισιόν και άλλων για την NSA. Διαβάσατε τα πρόσφατα ίσως σχόλια της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ, η οποία πιστεύει και διαβάζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ενδυνάμωση της Ευρώπης στον τομέα της συλλογής πληροφοριών και σύσφυξη των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ. Άρα μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι άλλο θα ακούσουμε κύριε Πρόεδρε. Εδώ δεν πρόκειται για την παραβίαση καμίας βασικής αρχής, απλώς για μια αγανάκτηση επειδή είπα έχουν περισσότερες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει ότι οι όλο και περισσότερες ενωσιακές δικαιοδοσίες έχει τελειώσει η περίοδος αυτή. Το αντίθετο ζητάει ο κόσμος τώρα. Η Ένωση να κάνει πολύ λιγότερα αλλά πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζίμερ έχει το λόγο. Um, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, Όταν μιλάμε για το, την τελευταία συνάντηση κορυφής, ε, πρέπει να πούμε ότι ήταν μια συνάντηση χαμένης ευκαιρίας. Αυτήν την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάστηκε στις πολιτικές ομάδες η ε, τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου. Και εκεί αναφέρεται ότι η εμπιστοσύνη στους ε, θεσμούς και η προθυμία προσέλευση εκλογές έχει μειωθεί ριζικά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που έγινε στο Συμβούλιο δεν βοηθάει στο να πάνε οι εκλογείς του χρόνου στις κάλπες για να αποφασίσουν ε, τι θέλουν να έχουν στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι πολιτική αποτυχία η οποία οφείλεται στις κυβερνήσεις ε, που ε, συμμετείχαν στο Συμβούλιο. Δεν έλαβαν καμία απόφαση για τα θέματα που σωρεύονται, που χρήζουν αποφάσεων, μετανάστευση, λαμπεντούζα, πολιτική ασύλου. Δεν βοήθησε και η Λαμπεντούζα στο να αμφισβητηθεί αυτή η πολιτική. Οι αρχηγοί της ε, Ιταλίας και της ε, Μάλτας ε, εστάλησαν απλά πίσω και προέκυψε μια δυσάρεστη κατάσταση διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και ανταυτού μας λένε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι τα αίτια στις χώρες της κρίσης να αρθούν τα αίτια αυτά και διαρωτώ. με εγώ η ε, κυβερνήσεις τι εννοούν ως αίτια ε, θα πρέπει ε, καταρχήν να δούνε λιγάκι τη συνέπεια που αναφέρεται ανάμεσα στην πολιτική συνέπειες και τις άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να δουν λιγάκι τους στόχους της χιλίτιας. Τίποτα δεν γίνεται. Και αν δεν τίθεται ούτε καν το βασικό θέμα και Πώς θα γίνουν όλα αυτά και πώς θα παρουσιαστούν αυτά ε, προς τα έξω, πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά και το πολιτές ε, νομικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ούτε καν δεν εξηγείται, εγώ διερωτώ με τότε τι γίνεται. Σε πάρα πολλά θέματα, εξακολουθούμε να είμαστε στην αρχή, ακούμε ότι η Μέρκελ και άλλοι εξακολουθούν να θέλουν να επιβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικά τους τα πρότυπα και δεν βλέπουμε να υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να πείσει τους νέους να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι δυνατόν να τα μετακυλίεται όλα αυτά σε εμά τους βουλευτές απλά και μόνο για να λέμε πόσο τέλεια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη στιγμή που ε, μένουν τόσα πολλά άλλη τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό. Και οι κυβερνήσεις ε, φέρνουν τεράστια ευθύνη και συνεχίζω να ερωτώ το πρόγραμμα για την Τραπεζική Ένωση. Μα όλοι γνωρίζουν ότι αν δεν γίνει κάτι σύντομα θα έχουμε ε, την επόμενη τραπεζική κρίση και είμαστε εξίσου ε, ελάχιστα προετοιμασμένη, όπως και σε αυτήν που προηγήθηκε. Τελικά τι θα γίνει. Δεν υπάρχει καμία σαφής δήλωση για το τι θα γίνει με αυτό το περίφημο Ταμείο Διάσωσης Τραπεζών. Ε, δεν υπάρχει καμία σαφής δήλωση για το ποιος θα πληρώνει τι, πότε, ποιος φέρει την ευθύνη. Όλα αυτά είναι ερωτήματα ε, που δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου και στην επόμενη συνάντηση κορφή απλά θα μας παρηγορήσετε και εμείς ως κοινοβούλιο μετά από δύο εβδομάδες θα ξαναπάρουμε το λόγο, θα κάνουμε τα σχόλιά μας ε, και αυτά, ποιος ασχολείται με αυτά, κανείς. Ε, έτσι κι αλλιώς αυτό που γίνεται σήμερα έχω την εντύπωση ότι απλά είναι υποχρεωτικό, αγκαρία είναι δηλαδή. Και τελικά μετά την τελευταία συνάντησή μας στο Στρασβούργο, τι έγινε. Εμείς υποβάλαμε τύπματα για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Θα μας πείτε τι θα γίνει με το 2013. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα το ότι ε, το έλλειμμα από 18 δις ε, ε, ορίζεται ευθύ εξ αρχή αυτή τη στιγμή και μας λένε ότι θα υπάρχει μια εμπροστοβαρής αντιμετώπιση για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας. Μιλάτε για την ψηφιακή Ευρώπη, όμως η χρηματοδότηση των προγραμμάτων είναι ανεπαρκής. Σε τελική ανάλυση είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ο τελευταίος οικονομολόγος γνωρίζει ότι όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν και εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει ε, να τα ξέραμε. Ελπίζω, Πρόεδρε, ε, να τα ξέρετε και απλά επειδή χτυπήσατε το σφυράκι φαντάζομαι ότι είναι απλά προς επιβεβαίωση αυτών που είπα εγώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τζίμ, ο κύριος Φάρατζ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Κύριε Βαντομπάη, και εδώ είχαμε να τα πούμε. 5 Νοεμβρίου είναι σήμερα, γιορτή στη Βρετανία. Πριν από 300 χρόνια έγινε μια προσπάθεια να καταστρέψουν ε, με δυναμή το κοινοβούλιο και να καταστρέψουν το σύνταγμά μας. Ε, Ευτυχώ απέτυχε και εσείς ε, με τις προσπάθειές σας να αντιμετωπίσετε τεχνοκρατικά τα πράγματα κάπως το ίδιο πράγμα προσπαθείτε να κάνετε. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ένωση τίποτα δεν γίνεται καλύτερο. 18 χρόνια στη σειρά, 19 τώρα μου λένε, δεν έχουν εγκριθεί ε, δεν έχει εγκριθεί ο απολογισμό. Όλα τα νούμερα ανάπτυξης που δίνεται, ένα πράγμα δεν μπορεί να ξεχάσετε, ότι η ανεργία των νέων στην ε, Μεσόγειο είναι πάνω από 50%. Και βεβαίως υπάρχει αύξηση της αντιπολίτευσης, της πραγματικής αντιπολίτευσης. Και όχι αναγκαστικά αντιπολίτευση την οποία θα ήθελα να μιλήσω εγώ. Σας ε, με κατηγόρησαν ε, πριν από λίγο καιρό ότι σας ρώτησα ποιος ήταν ο, ο ράφτης σας και πλήρωσε και τρία χιλιάρικα. Ε, μου απαντήσετε, ήταν νερό ε, στην πόλη. Το πρόβλημα είναι, ε, μεγάλωσε το ρούχο σας τα 3,5 χρόνια. Κανείς δεν μεγάλωσε στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό έχετε μια εκλογική θύελα. Κάτι δραματικό θα γίνει το Μάιο. Θα μπορούσατε να σταματήσετε αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις που θεωρείτε ότι μπαίνουν στο Κοινοβούλιο, αποδεχόμενοι ανοιχτά ότι ήρθε πλέον η ώρα να νομιμοποιήσετε με τον α ή τρόπο τα θεσμικά όργανα με ελεύθερα δημοψηφίσματα στα κράτη-μέλη για το αν θα έπρεπε εσείς να υπάρχετε. Οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί είπαν δεν πρέπει να υπάρχετε. Έβαλαν βέτο και όμως εκεί είστε κύριε Βανρομπάη. Έρχεται μια θύελα. Κάντε ό,τι μπορείτε για να νομιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αποφασίστε τουλάχιστον αν θέλετε να το κάνετε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Φάρατς. Ο, η κυρία Ο κύριος Στάντλερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Βαν Χομπέι, εγώ δεν συμμερίζομαι αυτά που είπατε και δεν είμαι μόνος. Ε, δεν συμφωνώ ότι έχει περάσει πλέον η οικονομική κρίση. Ε, απλά κερδίσατε και αγοράσατε ε, κάποιο χρόνο δαπανώντας δισεκατομμύρια. Τίποτα άλλο δεν καταφέρατε. Οι πολίτες όμως απαιτούν την σαφήνεια. Αναφέρομαι στα σημεία 43 και 44 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των κακών συσταγωγικά τραπεζών στο μέλλον θα χρησιμοποιούνται τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης. Και όχι κάποιο τυχαίος, ο κύριος Σόιμπλε ο ίδιος λέει και παραθέτω δεν θα χρησιμοποιηθούν χρήματα των φορολογουμένων για τη διάσωση των τραπεζών και πουδενή στα σίγουρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό μηχανισμό διάσωσης τέλος της παράθεσης. Ε, τώρα λοιπόν ε, κάνει και τη σύγκριση με την ε, S5 και λέει ότι εμείς είναι πλέον δεν θα δαπανίσουμε τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου για τις κακές τράπεζες. Και ρωτάμε αυτές τις κακές τράπεζες στα σημεία 43 και 44 αυτές πώς θα τις χρηματοδοτήσετε. Εδώ γίνεται λόγος για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης, κάτι που ο Σόιμπλε σε συμφωνία προφανώς με το Μαρκέλ και τον εταίρο της εταίρο του στην s τα αποκλείουν, τα αποκλείουν κατηγορηματικά. Και εμφανίστηκε η κυρία Λαγκάρτ που λέει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτεί το 1 δέκατο της φορολογίας σε όλες τις καταθέσεις. Αυτό είναι κατ' ουσίαν δίμευση. Είναι απαράδεκτο. Εμείς λοιπόν πριν από τις εκλογές απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφήνεια και ο πολίτης δικαιούται να μην του λένε συνέχεια ψέματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάω στο τρίτο, αυτή που επενείται την τραπεζική εποπτεία. Ποιοι ήταν οι κανόνες για αυτήν. Δεν υπάρχουν κανόνες, τους καταργήσατε τα υπόλοιπα των κανονισμών που υπήρχαν ε, καταργήθηκαν. Ποιοι κανόνες λοιπόν θα ισχύουν. Ε, κάποιοι λένε η Βασιλεία τρια μα δεν είναι αυτό ο κανόνας, δεν φτάνει ε, για τη ζούγκλα των κερδοσκόπων ή για να ελέγξει κανείς μια τράπεζα πρέπει να υπάρχει κάποιος κανονισμός το πώς χορηγούνται τα δάνεια. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες που ισχύουν υποτίθεται. Πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει το θάρρος να πει αυτοί είναι οι κανόνες που θα ισχύουν για τις τράπεζες και αυτοί οι κανόνες είναι απαραίτητοι. Πριν λοιπόν επιβληθεί η τραπεζική εποπτεία πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι δύο θέματα που δείχνουν ότι δεν επιλύσατε τίποτα απλά ε, σπαταλώντας τα δισεκατομμύρια του φορολογούμενου αγοράσατε χρόνο. Και ελπίζω γι' αυτό το λόγο θα σας τιμωρήσει ο πολίτης στις επόμενες εκλογές και θα έχει και δίκιο. Ωρα. Πάμε τώρα στις απαντήσεις ε, από την Επιτροπή. Ο Σεύκοβιτς έχει το λόγο. much, uh, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα συμφωνούσα με εκείνους τους ομιλητές που μας θύμεσαν ότι η ανάκαμψη είναι εύθευστη. Αυτό ήταν ε, σαφές και στην δήλωσή μου. Βλέπουμε ότι ήρθε η ανάκαμψη, αλλά είναι πολύ ευάλωτη. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Οι αγορές καθυστερούν ε, να πάρουν μπρος έξι μήνες και περισσότερο μετά την ανάκαμψη. Άρα πρέπει να συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, στερεώσουμε την ανάπτυξη και να ανταποκριθεί αυτό και σε αύξηση της απασχόλησης. Συμφωνώ και με εσάς που πιέζετε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα για τους νέους. Είναι σαφές ότι αναπτύξαμε και διαμορφώσαμε νέα εργαλεία. Με εξέπληξε ωστόσο όταν είδα πόσα κράτη-μέλη ήδη παρουσιάζουν και υλοποιούν προγράμματα εγγύησης νέων, ενώ έχουμε πάρει πληροφορίες μόνο από έξι κράτη-μέλη. Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να αναπτύξουν τα προγράμματα αυτά. Υπάρχουν κονδύλια της Ένωσης που θα καταμηθούν στο τομέα αυτό μέσω του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και που πρέπει να ξεκινήσουν ή δυνατόν και από πρώτου 14. Αν θέλουμε να διδαχθούμε από το παρελθόν και από τις εκκλήσεις της αγοράς εργασίας θα δίναμε έμφαση στα προσόντα που στερούμε. Θα έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο κενές θέσεις στο χώρο της ψηφιακής, των δραστηριοτήτων ψηφιακής, ε, ψηφι, ψηφιακής οικονομίας πρέπει να εισάγουμε, ενώ έχουμε μεγάλη ανεργία, πρέπει ταυτόχρονα να φέρουμε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Αυτή, αυτό το, πρέπει να συντεριάσουμε τις ε, ανάγκες με την προσφορά που υπάρχει. Τραπεζική Ένωση. Προφανώς είναι κρίσιμη η σύνοδος του Οκτωβρίου. Ήταν σημαντική, πολύ σημαντική, διότι πέρασε την ατμόσφαιρα της ανάγκης επίγουσας αντιμετώπισης του θέματος, τόσο ώστε το Δεκέμβριο να έχουμε έτοιμα όλα τα δημοσιονομικά εργαλεία και τα συστήματα μας για τον πλήρη ολοκληρωμένο έλεγχο που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στον τραπεζικό τομέα της Ένωσης του χρόνου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα... το τελευταίο κομμάτι του παζλ που πρέπει να φτιάξουμε για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρώπης και να αντιμετωπίσουμε τον φόβο που κάπως συνδέεται και με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Ελπίζω επίσης και ότι οι Υπουργοί Οικονομικών θα ακούσουν την έκκληση για επίγουσα δράση από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Στο θέμα της χρηματοδότησης, επαναλαμβάνω ότι ζητούμε από τα κράτη-μέλη να μας βοηθήσουν να πετύχουμε αυτή την κρίσιμη μάζα για την διαμόρφωση των δημοσιονομικών εργαλείων που θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε με ισχυρότερη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ιδίως με προσανατολισμό της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί και κάποια επιφυλακτικότητα από ορισμένα κράτη-μέλη για τα προγράμματα αυτά. Ελπίζουμε ωστόσο ότι μετά τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών κυβερνήσεων θα υπάρξει μεγαλύτερος ενθουσιασμός για το πρόγραμμα αυτό. Για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την ετήσια έκθεση ανάπτυξης, η Επιτροπή θα επανέλθει με τις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης ε, μέσα Νοεμβρίου. Ελπίζω ότι θα έχουμε διδαχθεί από τα πλήν και τα σύν του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα εξυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, προωθούμε την οικονομική διακυβέρνηση. Για τους προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014, ξέρετε, είναι λεπτό θέμα, ξέρετε πόσο δύσκολες είναι οι διαπραγματεύσεις, αλλά θα ήθελα να δείξω και κάποια αισιοδοξία από πλευράς Επιτροπής. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε φαντασία που έχουμε για να έχουμε δημιουργικές λύσεις με, και πιστεύω ότι με μια ουσιαστική πολιτική βούληση, θα καλύψουμε τα κενά, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και θα λυθεί το ζήτημα πολύ σύντομα. Για την προστασία δεδομένων και τις τηλεπικοινωνίες. Νομίζω εδώ τα πράγματα θα σαφή και πέρασε ένα σαφές μήνυμα και από την Επιτροπή. Η... Χρειάζεται αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας στις Ηνωμένε Πολιτείε. Επίσης, οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου πρέπει να συνεχιστεί. Δεν θεωρούμε ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών πρέπει να είναι ένα δώρο προς τη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν και δεν πρέπει να θεωρηθεί κάτι τέτοιο. Έχει πλονεκτήματα και για τις δύο πλευρές και χρειάζεται να διαπραγματευτούμε σκληρά για να υπερασπιστούμε τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης τομέα του εμπορίου, της τυποποίηση, ενώ ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε σε άλλο πλαίσιο να εξασφαλίσουμε ότι η προστασία δεδομένων θα επιτευχθεί. Κάτι που μπορεί να γίνει αν υπάρξει ενιαία θέση της Ένωσης σε αυτό το λεπτό θέμα. Για την τελευταία παρατήρηση του κυρίου Φαν Όντεν και τα σχόλιά του για τον διοικητικό φόρτο. Πρέπει να σας πω ότι πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έγινε μια συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής, του Πρωθυπουργού της Βρετανίας και μιας ομάδας ε, βιομηχάνων που καλωσόρισαν ιδιαίτερα τις νέες προτάσεις της Επιτροπής με το REFIT. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι βλέπουμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό και χρειαζόμαστε στέρεη συνεργασία και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου διότι πολλές προτάσεις μας για απλοποίηση βρίσκονται ακόμα στα τραπέζια πραγματεύσεων του Συμβουλίου και του, του Κοινοβουλίου. Για τις περικοπές στη διοίκηση τις κάναμε. Θα υπάρξει μια περικοπή 5%. Ταυτόχρονα οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δουλέψουν περισσότερο για τον ίδιο μισθό που είναι παγωμένος για πολλά χρόνια. Δεν θα ήθελα να συγκρίνω το μέγεθος της Επιτροπής με το μέγεθος ορισμένων Υπουργείων στη Βρετανία ιδίω που έχουν πάνω από δύο-τρεις δύο, φορές περισσότερους υπαλλήλους ε, από ότι η Κομισιόν. Ε, το Οικονομικών έχει 76.000 υπαλλήλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεύκοβιτς. Ο πρόεδρος κύριος Βαν Ρομπάιχ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάποιος είπε ότι δεν υπήρχαν εκπλήξεις σε αυτό το Συμβούλιο, αλλά και ορισμένες από τις αντιδράσεις εδώ μέσα ήταν χωρίς έκπληξη. Είχα την εντύπωση ότι τα έχω ξανακούσει όλα αυτά. Αν και η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει αλλάξει πολύ εδώ και ένα χρόνο. Πολύ. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει ορισμένους από εσά να ασκείτε πάντα την ίδια κριτική. Δεν ήμουν υπεραισιόδοξος, χρησιμοποίησα, δεν χρησιμοποίησα ούτε καν έναν φρόνιμο, μια φρόνιμη αισιοδοξία. Είπα απλώς ότι δημοσιονομικά η υπαρξιακή κρίση της Ευρωζώνης έχει λήξει. Αυτό όλοι το δέχονται. Αλλά βέβαια παραμένουν πολύ σοβαρά προβλήματα και η ασθένεια δεν έχει γιατρευτεί. Εδώ συμφωνώ. Γι' αυτό εργαζόμαστε τόσο σκληρά και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ορισμένοι λένε δεν έγινε τίποτα στο Συμβούλιο αυτό. Δεν ελήφθη καμία απόφαση, όλα έμειναν παγωμένα. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε πολύ ώρα για, το ψηφιακό πρόγραμμα, για την καινοτομία, καθώς και για την ενέργεια τον Μάιο και θα μιλήσουμε το ίδιο πολύ για την βιομηχανία της άμυνας και για την ανταγωνιστικότητα τον Φεβρουάριο. Αυτά είναι προγράμματα μέσω και πρόθεσμα που δεν ενδιαφέρουν πολλούς βέβαια αλλά που είναι ουσιώδη για το μέλλον. Και εδώ ελήφθησαν αποφάσεις. Σαφείς, βάλαμε ημερομηνίε, δημιουργήσαμε εργαλεία επεξεργαστήκαμε στρατηγική. Αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον και έγινε για πολλά θέματα σε πολλά συμβούλια κάτι τέτοιο. Αυτοί που λένε όλα είναι παγωμένα, δεν αποφασίστηκε τίποτα, αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Βράχει πρόθεσμα. Το θέμα της εξυγίανσης των τραπεζών ή της αντιμετώπισης των κρίσεων. Η Κομισιόν έχει κάνει μια πρόταση που ακόμα συζητιέται και θα αποφασίσει το Συμβούλιο το Δεκέμβριο σας διαβεβαιώνω φυσικά χρειάζεται χρειάζονται λίγοι μήνες για τόσο σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Θα έλεγα μάλιστα ότι κινούμαστε ιδιαίτερα γρήγορα. Στο τέλος του έτους θα έχει ληφθεί μια πολιτική απόφαση πέραν από την εποπτεία και γι' αυτό πριν από δύο χρόνια, και αυτό πριν από δύο χρόνια θα ήταν ανήκουστο. Αρχίσαμε τη συζήτηση τον Ιούνιο του 12, η πολιτική δουλειά τελείωσε τον Δεκέμβριο, πάλι Δεκέμβριο, και τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε και θα αποφασιστεί τελικά η ενιαία εποπτεία. Όταν τον περασμένο Ιούνιο σας είπα ότι έχει αποφασιστεί βασικά η δημιουργία ενός εργαλείου εποπτείας. Κανείς δεν με πίστεψε και τώρα υπάρχει. Το ίδιο θα γίνει και με την διευθέτηση των κρίσεων. Και ελπίζω όλα αυτά να τελειώσουν πριν λήξει η θητεία. Η πρόταση της Κομισιόν δεν λέω ότι θα γίνει δεκτή ως έχει, αλλά βασικά τράπεζες έχουν συμφωνήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από μερικούς μήνες επίσης τα έχει δεχτεί όλα αυτά τον Ιούνιο. Οι συμβατικές υποχρεώσεις είναι θέμα πολύπλοκο και είναι όμως απαραίτητο για το συντονισμό, κυρία Βόρτμαν Κόλ. Έγινε λόγος για τον οικονομικό συντονισμό, θα το αποφασίσουμε το Δεκέμβριο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι η συζήτηση ήταν ωφέλιμη και θα γίνει συγκεκριμένη πρόταση που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Και αν στην Τραπεζική Ένωση έχουμε την ενιαία εποπτεία, την επίλυση των κρίσεων για όλη την Ευρωζώνη και όσους θέλουν να μπουν σε αυτήν το μέλλον. Αν έχουμε επίσης τις συμβατικές αυτές διευθετήσεις, όλα αυτά μαζί με την Τραπεζική Ένωση, την Εξάμετρο και τη Δίμετρο βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της έκθεσης των τεσσάρων προέδρων θα έχει πραγματοποιηθεί. Και αυτό είναι ικανοποιητικό πριν λήξει η θητεία μου και της Κομισιόν καθώς και του Κοινοβουλίου να έχουμε συμπληρώσει τόσο σημαντική δουλειά. Σε σύγκριση ιδίω με ό,τι αναμενόταν πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη Λαμπεντούζα. Άκουσα τι είπε η κυρία Χάρμς ότι είναι σκάνδαλο κτλ. Αλλά ο βασικός ενδιαφερόμενος, ο Υπουργός Λέτα, είναι πολύ ικανοποιημένο από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχουν συμπεράσματα βράχη πρόθεσμα και το Δεκέμβριο το Συμβούλιο Υπουργών θα λάβει αποφάσεις, όχι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών, για τα πρόθεσμα αυτά θέματα, για την ενδυνάμωση του Frontex, για το Eurosur και άλλες πρωτοβουλίες εποπτείας και αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Όσο για τη διαμάχη, την πολεμική διαμάχη του καλοκαιριού με τις τελευταίες αποκαλύψεις πριν από μερικές εβδομάδες για τα κατασκοπευτικά και εδώ ο κύριος ενδιαφερόμενος, δηλαδή η Γερμανίδα Καγκελάριος, είναι πολύ, πολύ ικανοποιημένη από τα συμπεράσματα στα οποία συμμετέσχε. Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι λοιπόν, μαζί με άλλους, είναι αυτοί που έγραψαν αυτό το κείμενο. Πρέπει λοιπόν και εδώ να ξέρουμε τι λέμε. Ελπίζω να υπάρξει συμφωνία το Νοέμβριο για το Πουδουπού και για τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και όπως και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχω και εγώ απογοητευτεί γιατί σε επίπεδο κρατών μελών δεν έχει γίνει αρκετή πρόοδος για να υποβληθούν προγράμματα, αλλά αν εγκριθεί το που πριν το τέλος του έτους, μάλλον τον Νοέμβριο, ελπίζω τουλάχιστον, τότε μπορεί να αρχίσει η χρηματοδότηση ήδη από την 1η Ιανουαρίου. Με την ευθύνη βέβαια της Λιθουανικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελική συμφωνία. Και συμμερίζομαι αυτόν το, αυτή την μετριοπαθή αισιοδοξία που ανέφεραν ορισμένοι για την έγκριση του Πουδοπού. Τέλος, πριν από 3,5 χρόνια έλεγαν ότι έμοιαζα με τραπεζικό υπάλληλο. Τώρα από μόνος μου είμαι σε θέση να σταματήσω μία εκλογική θύελα. Ένας άνθρωπος δηλαδή μόνος του να έχει τη δυνατότητα να σταματήσει μια δίθεν εκλογική θύελα. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν δεν το λέγατε εσείς κύριε Φαράτζα, αλλά αφού το λέτε εσείς δεν με ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε τον ε, κύριο Βαν Χόμπεϊ και συνεχίζουμε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Στάντλα. Κοιτάξτε, ε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Να δούμε λιγάκι τι ακριβώς ε, θα είναι αυτή η Τραπεζική Ένωση. Δηλαδή, ποιου κανόνες ε, θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και ένας ευρωσκεπτικιστής ε, θα είχε να κερδίσει από κανόνες για, την, ε, για τις τράπεζες. Εσείς λέτε τώρα ότι έχετε θεσπίσει ένα μηχανισμό. Καλό αυτό. Ο εποπτική οργανισμό καλό είναι πάντα, αλλά ποια είναι τα κριτήρια που εφαρμόζουν αυτοί οι υπάλληλοι. κατά το δοκούν, λείπουν οι κανόνες και οι κανόνες αυτοί Ακόμα και σήμερα δεν μας το εξηγήσατε ποιοι είναι. Ο μηχανισμός ε, της ε, τραπεζικής εποπτείας ε, νομίζω ότι δεν καταρτώσατε τίποτα με αυτό, δυστυχώς ούτε και εμείς. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να φέρω. Το δεύτερο είναι ότι δεν επιφέρεται σαφήνεια με, σχετικά με το από πού θα προέλθουν τα κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλοποίηση των κακών τραπεζών. Και μάλιστα δεν λέτε και κατά πόσον στο μέλλον τις κακές τράπεζες θα τις αφήσετε να πτωχεύσουν. Αυτό θα ήταν είναι πιο λογικό. Οι μεγάλες αυτές ε, ανακοινώσεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν χρήματα προλογουμένων για τις κακές τράπεζες και αυτό πάλι λάθος είναι και λυπηρό και θα σας τιμωρήσει ο ε, ψηφοφόρος γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φαράζο έχει το λόγο. Θυμώσατε για ένα λεπτό, ξαφνικά πήρα, παθιάσατε, αυτό ήταν λαμπρό, να το κάνετε. Ο κύριος Βαν Ρομπάι που μιλούσε για τον ε, ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για το Ταμείο Εξυγίανσης. Ο κόσμος όμως μιλάει για κάτι άλλο, την έλλειψη δουλειάς, το άνοιγμα των αγορών ε, στους ε, πολίτες Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Ξέρετε τις θέσεις μου κύριε Βαν Ρομπάι για το δημοψήφισμα. Αν έρθετε και μου επιτεθείτε για αυτές τις θέσεις μου, ίσως να έχουμε πραγματικές ευρωεκλογέ. Δυστυχώς ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιείτε εσείς δεν είναι η γλώσσα των πολιτών. Κάθεστε με τη σημαία από πίσω σας. Λοιπόν, η σημαία αυτή απορρίφθηκε από τους Γάλλους, απορρίφθηκε από τους ε, Ολλανδούς το 2005. Δεν έχετε νομιμοποίηση, ελάτε να παλέψουμε το Μάιο. Ευχαριστούμε κύριε Φάρατζ. Η κυρία Τσίμερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης ε, και για τις ε, απαντήσεις που δόθησαν ε, τόσο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής όσο και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να συνεχίσω. Κύριε Σεύκοβιτς, εσείς επισημάνατε το ότι χαιρόσαστε πάρα πολύ για το γεγονός ότι ήδη έξι κράτη ε, έχουν καταβάλει τα απαραίτητα ποσά στο Ταμείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Αν όμως ισχύει αυτό ότι θέλουμε εμπροστοβαρή αντιμετώπιση για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα για τους νέους, τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η προσέγγιση σημαίνει ότι αυτά ε, που είχαμε από πέρυσι θα τα χρησιμοποιήσουμε εφέτος ε, για το 2014 και για το 2015 και αυτά που είχαν προσφερθεί για το 2014-2015 θα πάνε προς τα πίσω. Δηλαδή δεν προσθέθηκε δόθηκαν κονδύλια, απλά υπήρχε μία, υπήρξε μια διαφορετική κατανομή. Και τι είδους εγγύηση έχουμε για το ότι μετά το 2015 και το 2016 ε, το πρόγραμμα, το πρόγραμμα δεν θα αποτύχει. Ποιες είναι οι εγγύησεις που έχουμε για τη χρηματοδότηση άλλων σημαντικών ε, πρωτοβουλειών απασχόλησης, ε, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Μήπως αυτά χάσουν από χρηματοδότηση κατά τα επόμενα έτη, γιατί και αυτά είναι σημαντικά. Και να σας παραπέμψω και στην ιστορία με την Αμερικανική Υπηρεσία Ασφαλείας. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση στο ερώτημα τι ακριβώς ε, η υπηρεσία αυτή ε, και άλλες μυστικές υπηρεσίες και οι Βρετανικοί επέτρεψαν στον εαυτό τους ε, πρέπει να εστιατούμε στο εξή. η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να εμφανιστεί με σαφήνα και να πει δεν γίνεται αυτό δεν το επιτρέπουμε είναι πρόθυμα τα κράτη-μέλη να ε, προσφέρουν ας πούμε πολιτικό άσυλο στον κύριο Σνούντεν κοιτάξτε αυτά είναι ερωτήματα που περιμένουν οι νέοι να απαντηθούν ο κύριος Βανόρντεν έχει το λόγο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε κάτι που είπε ο κύριος Σεύκοβιτς θέλω να αναφερθώ. Βέβαια, η task force των επιχειρήσεων με συμμετοχή πρωθυπουργών και της Κομισιόν ήταν καλή, αλλά εμείς θέλουμε πραγματικά αποτελέσματα, δηλαδή αναστολή των νέων νομοθετημάτων, κατάργηση παλαιών νομοθετημάτων που είναι τμήμα του κεκτημένου και περικοπή του κόστους. Θέλουμε πραγματικά αποτελέσματα. Κάτι δηλαδή που και ο David Κάβερον και άλλοι ηγέτες θέλουν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναδώσει στα κράτη-μέλη ορισμένες δικαιοδοσίες έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα για το θέμα που ενδιαφέρει τους πάντες, δηλαδή την οικονομία. Δεν συμφωνούμε όλοι ότι τελείωσε η κρίση, εγώ φαντάζομαι ότι δεν τελείωσε ακόμη, αλλά ο βαθμός στον οποίο η Ένωση θα δεχτεί αποτελέσματα ενός πιθανού δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες θα δείξει που βρισκόμαστε, αν έχουν το θάρρος δηλαδή οι ηγέτες της Ευρώπης να, ρωτή, να ζητήσουν από τους πολίτες να απαντήσουν. Χάρμς. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι στη Μεγάλη Βρετανία πρέπει να συζητηθεί το ότι το μεγάλο βάρος ε, που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό οργανώνεται στο City του Λονδίνου και κοιτάξτε κάνετε πολύ μεγάλο λάθος το να περασπίσετε συνεχώς λάθος κανόνες αγοράς και να μπλοκάρετε την Τραπεζική Ένωση. Τώρα, κατά πόσον με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσετε μόνιμα θέσει απασχόληση στη Μεγάλη Βρετανία, πολύ το αμφιβάλλω, θα δούμε. Διάβασα σε μια εφημερίδα ότι ο κύριο Φάιμαν από την Αυστρία στο τέλο τη συνάντηση δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση τη Μέρκελ για εκείνον μάλλον δεν θα επιτύχει και εκείνος δεν είναι πρόθυμος ε, να υπογράφει συμβάσεις που επιβάλλονται εκβιαστικά και είπε επίσης ε, ότι τα κονδύλια για την ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί κανείς να τα πάρει μόνο εφόσον δεχτεί να υποκύψει σε μία μεταρρύθμιση που είναι όμως κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά διάβασα και το ότι εσείς εδώ δεν τα αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κάτι άλλο για τον κύριο Σνόντεν. Είπαμε, ο κύριος Σνόντεν είναι ήρωας. Είναι ο ήρωας πολλών νέων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι μέσω αυτού ξαναθυμούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποφασίζουν βέβαια να εφαρμόσουν κανόνες περί ασύλου και το γεγονός ότι δεν τα εξηγείται αυτά, δεν εξηγείται καν γιατί δεν του προσφέρετε άσυλο. Ένας λόγος είναι γιατί δεν μπορείτε να τον προστατεύσετε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και με αυτό δεν ενθαρρύνει κανείς τους νέους να στηρίξουν την ευρωπαϊκή ιδέα. Παρμπάνοβα. Πρόεδρε. οι ανισότητες είναι αυτή τη στιγμή το βασικό θέμα στην Ευρώπη. Αυξάνεται η ξενοφοβία και αυτό δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες. Πρέπει να είσαστε πιο δυνατοί και πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά σας. Του χρόνου έχουμε εκλογές. Το κοινοβούλιο, το σώμα θα, θα εμφανιστεί ενώπιον των ψηφοφόρων. Και εσείς μας μπλοκάρετε. Δεν κατεβαίνετε στις εκλογές, κατεβαίνουμε εμείς. Εμάς θα μας κρίνουν. Και εμείς πιστεύουμε ότι η, η λύση είναι μεγα, περισσότερη Ευρώπη, μεγαλύτερη συνοχή. Δεν είμαστε επαρκώς έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους Αμερικανούς, τους Κινέζους, τους Ινδούς. Ο ίδιος ο Ομπάμα έχει αρχίσει να λέει ότι δεν είμαστε πλέον στρατηγική εταίροι των ΗΠΑ ταν πέρα από μας, την Κίνα, την Ινδία και είπαν, το είπαν πολύ σαφέ, σαφώς πριν από δύο χρόνια που είχαμε συναντήσει η ομάδα μας στην ε, κυβέρνηση Ομπάμα και μας είπαν, Ομπάμα, και μας είπαν σαφώς ότι και στη Γερουσία και στη Βουλή η οικονομική κρίση δεν είναι αποτέλεσμα πλέον της κρίσης της ΕΠΑ, αλλά είναι καθαρή κρίση του τρόπου λήψης αποφάσεων στην Ένωση και της ίδιας της Ένωσης. Και εσείς είστε υπεύθυνοι που συνεχίζεται η κρίση. Πρέπει να είσαστε πιο ανοιχτοί στο να καταλαβαίνετε τι λύσεις θέλει ο κόσμος. Ευχαριστώ. Κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ. Κύριε Βανορόμπαρη σε μια απάντηση που προφανώς ε, απευθύνονταν σε μένα, είπατε ότι η παρέμβασή μου δεν ήταν έκπληξη. Και τονίσατε ότι τα τελευταία χρόνια άλλαξε το Συμβούλιο, ενώ οι σοσιαλιστές μένουν οι ίδιοι. Αυτό τι σημαίνει. Κατά με σημαίνει ότι η σοσιαλιστική ομάδα παραμένει η ίδια, ενώ το Συμβούλιο παρότι αλλάζει σε πρόσωπα, δεν αλλάζει σε στάση. Ωστόσο, δεν είναι αντίθετα με αυτά που θέλουμε όλα όσα κάνει το Συμβούλιο. Σε κάποια στοιχεία έχουμε διαφοροποιήσεις και σε κάποια έχουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία σε σχέση με αυτά που ε, εντοπίζει το Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε το τι μπορεί να πετύχει ο πρόεδρος του Συμβουλίου με το τι μπορεί να πετύχουν τα κράτη-μέλη. Η κριτική λοιπόν εν μέρη της παρέμβασής μου δεν αφορά εσάς, αφορά τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη που δεν ήταν ικανά σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση να δώσουν περισσότερα κονδύλια και ηλική υποδομή στις δύο ευρωπαϊκές υπηρεσίε που χρειάζεται να απαντήσουν στο θέμα αυτό, την, το ΕΑΖΟ και το Frontex. Είναι γεγονός ότι τον Ιούνιο θα υπάρχουν κάποιες στρατηγικές ε, καθευθυντήριες γραμμές. Συμφωνώ. Πιστεύω ότι η Ένωση χρειάζεται μια μεταναστευτική στρατηγική. Τριάμιση λεπτά. Χρειάζεται. Τρισήμιση λεπτά μου δώσετε πρόεδρε. Χρειάζεται έλεγα μια στρατηγική για τη μετανάστευση και η στρατηγική αυτή για τη μετανάστευση πρέπει να βασίζεται κατά βάση στην πρόληψη την συμφωνία με τις χώρες προέλευσης, την μείωση της φτώχειας, την βοήθεια στη μείωση της φτώχειας στις χώρες αυτές. Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή μερίσια διάταξη, η ομάδα μου συμμερίζεται εν γέννη τις θέσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο, παρότι πιστεύει ότι αυτή η στο πλαίσιο αυτής της μεγαλύτερης φιλοδοξίας που ανέφερε, ότι τα κράτη στο Συμβούλιο θα έπρεπε να πάνε παραπέρα. Δηλαδή, η ευρυζωνική ε, η ευρυζωνικότητα που συνδέεται με το Connecting Europe Facility που ωστόσο μειώθηκαν τα κονδύλια από τα 9 στα 1 δις. Σημαντική μείωση. Για την ε, τεχνολογία 4G. Η θέση της Ευρώπης είναι ε, αστεία σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 80% έχουν πρόσβαση, στην Ευρώπη 75% δεν έχουν πρόσβαση. Στον, εν ώψη του ορίζοντα 2020 το Κοινοβούλιο ζήτησε 103. Η, η Επιτροπή είπε 80 δις και τελικά θα είναι 70 στον προπολογισμό της Ένωσης. Τώρα για τους νέους. Μίλησε ο Αντιπρόεδρος για το ότι έξι μόνο χώρες ενέκριναν ήδη την στρατηγική απασχόληση των νέων. Αυτό είναι ένα στρατηγικό θέμα για την Ένωση και για την Ευρώπη. Οι νέοι χρειάζονται αποτελέσματα και αξίες. Και το μιλάει κανείς για αξίες, η πιο ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της Ένωσης, το Εράσμους, κινδυνεύει πραγματικά να εξαφανιστεί λόγω προσπαθειών της ίδιας της Ένωσης και κάποιων κρατών μελών της Ισπανίας στη συγκεκριμένη περίπτωση που απέσυραν την εθνική συνεισφορά στους ε, ερασμιακούς υπότροφους όταν, πηγαίνουν στις, όταν πήγαιναν στις χώρες που ήθελαν να πάνε. Ευχαριστώ κύριε Γκερέρο. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ως τελευταία ομιλήτρια θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Ακούσαμε πολλές επικρίσεις για πολλά θέματα που συζήτησε το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος Βαν Ρομπουή. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι την κρίση δεν μπορούμε να τη σβήσουμε απλώς. Για να λυθεί η κρίση χρειάζεται αλληλεγγύη και ευθύνη για να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αν δούμε τι πετύχαμε τον τελευταίο χρόνο, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ενίσχυση των θεσμών και έγκριση και εμβάθυνση της νομισματικής ένωσης. Επίσης, βασικό θεμέλιο παρέμεινε η ενωσιακή μέθοδος. Αλλά θα ήθελα να καλέσω τώρα το Συμβούλιο και την Κομισιόν να επενδύσουν περισσότερο στην αξιοπιστία αυτού του συστήματος που από κοινού δεχτήκαμε. Ανησυχώ ότι σε κάποιο πρόσεχες Συμβούλιο θα εγκριθούν διακυβερνητικά εργαλεία που θα υπονομεύσουν αυτή την αξιοπιστία αυτού του συστήματος. Παρακαλώ λοιπόν και εσάς να επιμείνετε στο από κοινού συμφωνηθέν σύστημα. Όσο βγαίνουμε από την κρίση πρέπει να επενδύσουμε σε μακροπρόθεσμα θέματα όπως την ψηφιακή αγορά ή το ενεργειακό που θα μπορούσε να είναι η επόμενη κρίση και πρέπει να το δούμε από τώρα κατά πολέμηση του προστατευτισμού, το refit και σημαντικά θέματα όπως την παράνομη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική. Πρόεδρε Βαν Ρόμπα, ούτε εγώ μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλά θα ήθελα να πω τα εξή. Σε δύο χρόνια είμαι σίγουροι ότι ως πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα θεωρηθείτε ως κάποιος που κατάφερε τα αδύνατα. Γιατί αν δούμε τι θεωρούνταν αδύνατο πριν από ένα-δύο χρόνια, διαπιστώνουμε ότι το αδύνατο δίθεν αυτό έχει εφαρμοστεί. Και ελπίζω να μπορούμε να έχουμε την εμπιστοσύνη σας και γι' αυτό. Ευχαριστώ τους πάντες και τον κύριο Βανερόμπου και τον αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς και καλή συνέχεια.